Thank you. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Είναι τιμή για μένα να είμαι εδώ ενώπιό σα σήμερα ω υποψήφια επίτροπο για την εσωτερική αγορά, βιομηχανία, μικρομεσαίε επιχειρήσει και επιχειρηματικότητα. Ελπίζω να μπορέσω να κερδίσω την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή σα για την αποστολή που μου εμπιστεύτηκε ο πρόεδρο Γιούγκερ. Μετά την οικονομική κρίση των τελευταίων έξι ετών υπάρχουν ορατά σημάδια ανάκαμψη. Όμω, ξακολουθούμε να χρειαζόμαστε κατεπηγόντω ανάπτυξη και απασχόληση. Και η Ευρώπη πρέπει να ξαναβρει το δρόμο προ την ευημερία, τον οικονομικό δυναμισμό και την κοινωνική συνοχή. Για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς, εγώ προσωπικά θέλω να εστιάσουμε στην πραγματική οικονομία, που πιστεύω ότι πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά του οικονομικού θεματολογίου της Ευρώπης. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Σίγουρα όχι επανερχόμενοι σε μια συζήτηση για το κατά πόσο χρειαζόμαστε μια Ευρώπη πιο φιλελεύθερη, πιο κοινωνική. Και τα δύο χρειαζόμαστε και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά συστατικά της Ευρώπης. Η ιστορική αγορά μπορεί να δώσει πολύ περισσότερα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις επιχειρήσεις μας όταν τις κάνει προτεραιότητα. Επίσης μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, διότι οι σύγχρονες οικονομίες βασίζονται σε αλυσίδες οικονομικών αξιών, όπου τα αγαθά, οι υπηρεσίες αλληλεξαρτώνται το ένα από το άλλο και όπου δεν υπάρχουν ε, ε, δίπλα μόνο οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη, αλλά μπορεί να είναι και πέραν των συνόρων. Θα συνεργαστώ με τους, ε, μάλλον θα συνεχίσω το έργο των προκατόχων μου Μπανιέτα Γιάννη και Νέλη Φερότση στην αποστολή μου και θα εστιάσω σε τέσσερις στόχους. Ανάπτυξη του πλήρους δυναμικού της εσωτερικής αγοράς, προώθηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας μέσω των επενδύσεων και της καινοτομία, αποδέσμευση απελευθέρωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στήριξη των ΜΜΕ και τέλο, ε, προώθηση της εσωτερική αγοράς πέραν των συνόρων μα. Θα αναφερθώ εν συντομή και στους τέσσερις αυτούς στόχους. Πρώτος στόχος ε, για την εστερική αγορά. Ε, έχετε ακούσει άπειρες φορές ότι η εστερική αγορά είναι το πλέον ε, σημαντικό εργαλείο που διαθέτουμε για τις θέσει εργασία και την ανάπτυξη. Όμως υπάρχουν ακόμη εμπόδια, υπάρχουν φραγμοί ή ξαναδημιουργούνται και αυτό είναι και ένα από τα συμπεράσματα της πρόσφατης μελέτης για το κόστος της μη Ευρώπης. Πρέπει να εστιάσουμε σε τομείς και περιοχές που έχουν το μεγαλύτερο αναπτυξιακό δυναμικό. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι παραμένουν σημαντικά εμπόδια για μια πλήρως ανεπτυγμένη αγορά υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι και νομικά και πρακτικά τα εμπόδια αυτά και πρέπει να τα ξεπεράσουμε, να βρούμε τρόπους να δημιουργήσουμε περισσότερη ανάπτυξη, για παράδειγμα μέσω της περαιτέρω χρήσης της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης θα πρέπει να εστιάσουμε σε τομείς που έχουν ξεκάθαρη σχέση με την βιομηχανική μας πολιτική και την πολιτική για τις ΜΜΕ. Παράδειγματο χάρη, επιχειρηματικές υπηρεσίες, σκευαστικός κλάδος, λιανικές πωλήσει. Επίσης, η εσωτερική αγορά των αγαθών, των εμπορευμάτων, έχει προχωρήσει ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, όμως σήμερα η διάκριση μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών δεν είναι τόσο σαφής πια. Γι' αυτό χρειάζεται απλούστευση και ενοποίηση της προσέγγισης που έχουμε ε, και για τα δύο σκέλη, προϊόντα και υπηρεσίες δηλαδή στην εσωτερική αγορά, τουλάχιστον σε ορισμένους τομείς. Επίσης θα ήθελα σε αυτό το πλαίσιο να αναφέρω την ενιαία ψηφιακή αγορά. Καιρός πια είναι αυτά τα πανταχού παρόντα ευφυή τηλέφωνα, smartphones, να τα συντεριάξουμε με ευφυείς πολιτικές, smart policies. Πρέπει να παγιώσουμε αλλά και να προωθήσουμε τα ίδια επιτευθέντα και γι' αυτό η αποτελεσματική εφαρμογή θα είναι προτεραιότητά μου. Όλοι οι κανόνες να εφαρμόζονται σωστά επί τόπου, με απλό, έγκαιρο, αποτελεσματικό τρόπο. Η διακυβέρνηση της εσωτερικής αγοράς ε, θα είναι το ίδιο σημαντική για εμένα όσο είναι για εσάς και θα διαδραματίσει πλήρη ρόλο στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τα κράτη-μέλη. Θα ζητήσω από τις υπηρεσίες μου να αξιοποιήσουν πλήρως τα εφιστάμενα εργαλεία για την αξιολόγηση του κόστους και ωφέλους της νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων αξιολογήσει αντικτύπου, τεστ για τις ΜΜΕ, ανταγωνιστικότητα εκ των υστέρων αξιολογήσεις κτλ. Με τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς που είναι αρμόδιος για την καλύτερη ρύθμιση και το REFIT θα συνεργαστώ πολύ στενά ώστε αυτά να ε, αντικατοπτρίζονται και σε όλες τις πρωτοβουλίες της Κομισιόν. Και βέβαια Τέλος, εξίσου σημαντικό όμως, ε, που είναι κινητήριο Μοχλό για την ανάπτυξη. Πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στου πολίτε μα, ότι η Ευρώπη είναι εκεί για αυτού. η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι στην υπηρεσία του. Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται λοιπόν κοινωνική διάσταση και γι' αυτό το σημείο θέλω να ξεκαθαρίσω απόλυτα το εξή. Δεν συμφωνώ με όσου υποστηρίζουν ότι η εσωτερική αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει διότι οι οικονομικές ελευθερίες δεν μπορούν να συμφιλειωθούν με τα κοινωνικά δικαιώματα ή τούμπαλιν. Φυσικά και υπάρχουν λεπτές ισορροπίες που πρέπει να βρεθούν. Ωστόσο δεν αμφιβάλλω σε καμία περίπτωση ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια εσωτερική αγορά η οποία θα βασίζεται στο κράτος δικαίου και θα λειτουργεί, θα λειτουργεί στην πράξη. Τούτου λεχθέντος ε, θέλω να τονίσω το προσωπικό μου ενδιαφέρον προς την κοινωνική επιχειρηματικότητα, που μπορεί πάρα πολύ καλά να συνδυάσει καινοτόμε λύσεις στα κοινωνικά προβλήματα. Με πεπισμένη ότι αν θέλουμε λύσεις μπορούμε να τις βρούμε, για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Επαγγελματικό Επισκεπτήριο που θα κάνει πολύ πιο εύκολο ε, το να βρει κανείς ε, να μπορεί κανείς να εργαστεί σε οποιοδήποτε άλλο μέσο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να σας ε, αναφέρω λίγα παραδείγματα που θα με απασχολήσουν κατά προτεραιότητα τους επόμενους μήνες. Πρώτα απ' όλα, πλήρη υλοποίηση της αγοράς για τις υπηρεσίες, μαζί με μια νέα στρατηγική για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Επίσης, το πακέτο για την προστασία των προϊόντων και την επιτήρηση της αγοράς η αποτελεσματική εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τις δημόσιες προμήθειες και η ενοποίηση του πλαισίου μας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η δεύτερη μεγάλη προτεραιότητα θα είναι η πρόθεση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας μέσω επενδύσεων και καινοτομίας. Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς μια στέρεη βιομηχανική βάση. Η βιομηχανία αντιπροσωπεύει τα τρία τέταρτα της έρευνας και καινοτομίας του ιδιωτικού τομέα στην Ένωση και τα τρία τέταρτα των εξαγωγών της Ευρώπης ε, με απόδοση 1 δισεκατομμύριο εμπορικό απόδο, ε, πλεόνασμα καθημερινά. Είναι η βιομηχανία και στην καρδιά της πραγματικής οικονομίας και πηγή ε, της δραστηριότητας ε, του τομέα των υπηρεσιών. Αλληλοεξαρτώμενα κατά συνέπεια τα εμπορεύματα και οι υπηρεσίες. Αν θέλει η Ευρώπη να είναι ευημερής, να ευημερήσει, να είναι ανταγωνιστική, ε, προηγμένη τεχνολογικά και βιώσιμη περιβαλλοντικά, πρέπει να προωθήσουμε την, την βιομηχανική της ανταγωνιστικότητα και μέχρι το 2020 ε, το οικονομικό βάρος της να φτάσει στο 20% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέσσερις είναι βασικής τομείς στη στρατηγική μου για τη βιομηχανία. Πρώτον, πρέπει η βιομηχανία να έχει προσιτή πρόσβαση ε, σε ενέργεια, ε, πρώτε ύλε, δεξιότητες. Είναι οι πιο υψηλέ ε, τιμές ενέργειας αυτές που έχουμε εδώ στην Ευρώπη σε σχέση με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Εξαρτώμαστε από εισαγωγέ μας για ενέργεια και για σημαντικές πρώτε ύλε και αυτό είναι πολύ σημαντικό για ενεργοβόρες βιομηχανίε που όμω πρέπει να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητά του. Θα προσπαθήσω να διευκολύνω περαιτέρω βελτιώσω τον τομέα της ενεργικής απόδοσης και να δείξω ότι συμβαθίζουν χέρι-χέρι η ανταγωνιστικότητα με τη βιωσιμότητα. Θα στηρίξω την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Θα συνεργαστώ με την συνάδελφό μου Μαριάν Τίσεν σε μια φιλόδοξη προσπάθεια να πληρώσουμε τα κενά δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για τις επιχειρήσεις όπως είναι τεχνολογία ή τα, έργα μηχανικού. Θα προωθήσω την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση όπως και την επιμόρφωση. Δεύτερον, το μεγαλύτερο πρόβλημα που μετωπίζει η μηχανία στην Ευρώπη είναι η δραματική μείωση των επενδύσεων που είναι 20% κάτω των επιπέδων πρώτης κρίσης. Θα στηρίξω σε αυτό το πλαίσιο τον Αντιπρόεδρο Κατάινεν ε, για να κινητοποιήσουμε ε, το πακέτο επενδύσεων του ύψους των 300 δις που θα προτείνει και πρέπει να φροντίσουμε να δαπανηθούν παραγωγικά οι πόροι αυτοί. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν όλη την εμπειρία που έχω με την περιφερειακή χρηματοδότηση ώστε οι επενδύσεις πραγματικά να βοηθήσουν ε, στην ε, ανοικοδόμηση του βιομηχανικού ιστού της Ευρώπης με την ε, στρατηγική μας για την ευφυή εξειδίκευση. Τέτον, η βιομηχανία Τρίτον, η βιομηχανία πρέπει να είναι σε θέση να επενδύσει στην καινοτομία και στον εξυγχρονισμό. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον φιλικό προ την καινοτομία. Οι ιδέε δηλαδή να στηρίζονται από τη σύλληψή του μέχρι την ώρα που θα εφαρμοστούν στην αγορά. Θα αξιοποιήσω όλα τα εργαλεία πολιτική που έχουμε στη διάθεσή μα. Από τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία, τη σχετική υποδομή για τη στήριξη ε, της ε, καινοτομίας και των τεχνολογιών μέσω της χρηματοδότησης ε, και της πολιτικής νοσίων συμβάσεων. Μαζί με τον συνάδελφο Κάρλος Μοέδας θέλω να αξιοποιήσω το πρόγραμμα Horizon 2020 και άλλα εργαλεία πολιτικής της Ένωσης για να στηρίξουμε τη βιομηχανική καινοτομία και σημαντικές τεχνολογίες όπως είναι η ψηφιακή, η βιοτεχνολογία, η νανοτεχνολογία, μεταποίηση κτλ. Τέταρτον, θα δώσω ιδιαίτερη προσοχή στι στρατηγικέ βιομηχανίε τη Ευρώπη. και θα ήθελα να σα αναφέρω κάποιου μεμονωμένου τομεί Στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδρομολογήσουμε τη διαδικασία CARS 2020, να αναθεωρήσουμε το πλαίσιο έγκριση τύπου και να δώσουμε μια ισχυρή όθηση στην παγκόσμια εναρμόνιση τη νομοθεσία ε, για τα αυτοκίνητα. Στον τομέα των χημικών, μαζί με τον συνάδελφο Καρμένου Βέλα, θα ε, προσπαθήσω και εγώ να βελτιώσουμε την υλοποίηση του REACH, ιδίω ό,τι αφορά τη διαδικασία για την χωρίση άδεια κυκλοφορίας. Στον τομέα της άμυνας θα εστιάσω στην εσωτερική αγορά, ε, στις διαγωνισμούς ε, για, αμυντικά, για αμυντικούς εξοπλισμούς, στον εξορθολογισμό των επενδύσεων με βάση τον οδικό χάρτη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στον κατασκευαστικό κλάδο θα ήθελα να γίνει ένας έλεγχος ε, της καταλληλότητας του τομέα και ανάλυση της υλοποίησης του κανονισμού για τα κατασκευαστικά για τα δομικά προϊόντα. Να είναι σαφές όμως ότι η προσέγγιση μου θα είναι συνολική, σφαιρική, θα εμπεριέχει όλους τους τομείς. Από τη χαλιβουργία μέχρι τον τουρισμό και τις δημιουργικέ βιομηχανίες λαμβάνοντας όμως υπόψη τι ιδιαιτερότητε του κάθε τομέα. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι επίση σαφέ ότι συνεργαζόμενοι με τους ε, βιομηχανικούς κλάδους ε, θα ε, ασχοληθώ με ιδιαίτερη προσοχή με τομείς που ενδιαφέρουν τους πολίτες. Πρώτον, στον τομέα των, ε, των υγειονομικών. Η εγγύηση της υγείας των ασθενών μας και των πολιτών μας να είστε βέβαιοι ότι θα είναι η βασική μου μέρημνα. Η υγεία και η ασφάλεια έρχονται πρώτα για μένα και προτίθεμαι να συνεργαστώ στενά για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την υγεία με τον συνάδελφο Βιτένης της τον υποψήφιο για την υγεία επίτροπο. Δεύτερον, η βιομηχανία μας πρέπει να παραμείνει βιώσιμη. Πρέπει επίσης να δώσουμε προσοχή και στους όρους για την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας. Εξού και προτίθεμαι να εξετάσω το ενδεχόμενο πρόθεση ενός πακέτου μέτρων που θα προωθούν τις καθαρές τεχνολογίες και μια προσέγγιση για την αποδοτική και βασιζόμενη στην αγορά χρήση των πόρων. Το 2015 θα προτείνω ένα πλήρω δικό χάρτη με όλες τις δράσεις για τη στήριξη της βιομηχανίας και θα βάλω την ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 και στο κέντρο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τρίτη προτεραιότητα, ΜΜΕ. Όλες οι εταιρείες χρειάζονται ένα ε, φιλικό ε, για ε, την επιχειρηματικότητα ρυθμιστικό πλαίσιο. Θα επιμείνω στην απλούστευση και την προβλεψιμότητα για τι επιχειρήσει και θα δώσω ιδιαίτερη προσοχή στι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Θα αξιοποιήσω πλήρω τα 2,3 δισεκατομμύρια του προγράμματο COSME, ιδίω για τη στήριξη τη πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και για την αναβάθμιση του δικτύου Enterprise Europe, ώστε να μπορούν οι ΜΜΕ να αντλούν τα μέγιστα δυνατά ωφέλη από την εσωτερική αγορά και να μπορούν να βρίσκουν αγορέ στο εξωτερικό. Όλε οι πρωτοβουλίε που προτείνω θα υποβληθούν στο λεγόμενο τεστ ΜΜΕ ε, σε μια δοκιμή δοκιμή ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να μην επηρεάζονται δυσανάλογα οι μικρότερες εταιρείες. Επίσης προτείνω ε, να έχουμε ε, μια αναθεωρημένη Small Business Act για την Ευρώπη με στόχο οπουδήποτε στην Ευρώπη να μειωθούν δραστικά τα έξοδα και το κόστος για την σύσταση μιας επιχείρησης και να είναι πολύ πιο εύκολη και γρήγορη η διαδικασία αδειοδότης. Πρέπει επίσης να μειώσουμε το διοικητικό άχθος, να έχουμε ηλεκτρονικές μοναπευθυντικές θηρίδες, ε, να διευκολύνουμε τις μεταφορές, ε, ε, τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων. Επίσης προτείνω διευκόλυνση της διαχείρισης δίκαιης δίκαιων υποθέσεων ή ειλικρινών υποθέσεων χρεοκοπίας, ώστε οι ειλικρινείς επιχειρηματίες να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία και θα συνεργαστώ με την Επίτροπο, την κυρία Γιούροβα, που είναι αρμόδια για τα θέματα δικαιοσύνη. Τέταρτη προτεραιότητα, πώ θα προωθήσουμε την εσωτερική αγορά πέραν των ε, συνόρων. Σίγουρα βασίζεται η μελλοντική μα ευημερία στι διεθνεί αγορέ. Η οικονομία τη Ευρώπη χρειάζεται πρόσβαση σε αγορέ και εντό Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίω. Θα συνεργαστώ λοιπόν με, τον, με την αρμόδια για το εμπόριο Επίτροπο, την κυρία Σεσίλια Μάλμστρομ, για να στηρίξουμε το άνοιγμα των αγορών εκτό τη Ευρώπη σε πνεύμα αμοιβαιότητα και αμοιβαίου ωφέλου. Ιδιαίτερα σκέφτομαι τις ΗΠΑ Πολιτείε και την Ιαπωνία, όπου έχουμε ήδη ε, σε εξέλιξη τις διαπραγματεύσεις. Πρέπει και από τις δύο πλευρές να γίνει μείωση των ε, δασμών ε, και των, άρση των μη δασμολογικών φραγμών, να έχουμε ανοιχτέ υπηρεσίε αγορών και βελτιωμένη πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα για τις διάφορες δημόσιες προμήθειες. Αλλά ταυτόχρονα, όπως και ο πρόεδρος Γιούγκερ, δεν μπορεί και δεν θα γίνει αυτό σε βάρος των προτύπων μας και των κανόνων μας. Βέβαια θα δώσουμε προσοχή και σε αναδυόμενες αγορές όπως είναι η Κίνα ή χώρες από ε, την ε, γειτονιά μας. Άλλη μια πρόταση, άλλη μια πρόταση, μου επιτρέπετε. Βεβαίως, βεβαίως λέει ο κύριος Μπούζεκ. Ξέρετε, κάποιες φορές στην Ένωση υπάρχει η εντύπωση ότι ό,τι κάνουμε για την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς ε, γίνεται μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό είναι λάθος. Λάθος αντίληψη. Η εσωτερική αγορά για μένα είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Είναι το θεμέλιο της ευρωπαϊκής μας οικονομίας και επηρεάζει κάθε μεμονωμένη εταιρεία, κάθε μεμονωμένη επιχείρηση. Έξω και η εσωτερική αγορά από κοινού με την καινοτομία θα πρέπει να δώσει αποτελέσματα για να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δημιουργώντας την τόσο απαραίτητη ανάπτυξη και θέση εργασία στους πολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ. Ας ξαναβάλουμε την Ευρώπη μπροστά. Ας αρχίσουμε δουλειά. Ευχαριστώ.